Στην ε, Ευρωζώνη και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, ανάκαμψη στην αγορά In this budget... απασχόλησης. Σε αυτό το προλογισμό... Σε προπολογισμό εργαστήκαμε πολύ σκληρά προκειμένου να στηρίξουμε τις δράσεις της Ευρωπαϊκής ε, και να αντιμετωπίσουμε τις νέες ε, προκλήσεις, ιδιαίτερα αυτές που προέκυψαν στη γειτονική μας περιοχή, στην Ουκρανία, τη Συρία, το Ιράκ, για να αναφέρουμε ορισμένε από αυτές, και τον αντίκτυπο που έχει αυτή η αστάθεια στη μετανάστευση. Γιατί όταν είχαμε τη συζήτηση για το σχέδιο πληρωμών, διαπιστώσαμε ότι οι εξωτερικές δράσεις, ότι και τις εξωτερικές δράσεις ε, οι πιστώσεις πληρωμών ήταν σε δραματική κατάσταση και για το 2016 το αντιμετωπίζουμε. Έχουμε 28% αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για τι εξωτερικέ δράσεις και 36% αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για τη μετανάστευση. Θα επανέλθω στα σημεία αυτά όταν επισέλθουμε στις λεπτομέρειες του προπολογισμού. Και τελευταίο σημείο εξίσου σημαντικό, το αναφέρατε και στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και ε, δικαίως, στο σχέδιο προπολογισμού του 2016 συμπεριλάβαμε και τη συμφωνία για το σχέδιο πληρωμών, προκειμένου να μειώσουμε τους ανεξόφλητους λογαριασμούς το 2016 και να τους φέρουμε στο στόχο που περιλαμβάνει η συμφωνία των πληρωμών, δηλαδή στα 2 δισεκατομμύρια. Και περιλάβαμε το 21,1 δισεκατομμύρια, ιδιαίτερα για να μειώσουμε τις, τους απλήρωτους λογαριασμούς. Ποια είναι τα βασικά σημεία του νέου προπολογισμού, ό,τι αφορά τις την ανάληψη υποχρεώσεων έχουμε 153,5 δισεκατομμύρια, 1,04% του ευρωπαϊκού ΑΕ. Και αν εξουδετερώσουμε το, την, τον προγραμματισμό των αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2015, θα οδηγηθούμε σε ελαφριά αύξηση 2,4%. Αν όμως δεν κάνουμε αυτή την προσπάθεια, θα έχουμε πιθανότητα μείωσης. Γιατί 21 δισεκατομμύρια των αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν τηρήθηκαν θα πρέπει να τις μετακυλήσουμε στον προϋπολογισμό του 2015. Έχουμε ένα άνετο περιθώριο, 2,2 δισεκατομμύρια στις αναλήψεις υποχρεώσεων. Χρησιμοποιούμε το γενικό ε, περιθώριο των ε, αναλήψεων υποχρεώσεων, 351,4 εκατομμύρια και το μηχανισμό ευελιξίας 124 εκατομμύρια για τις πληρωμές. Έχουμε καλύτερο προϋπολογισμό φέτος από την πέρυσι. 143,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή 0,98% του Ευρωπαϊκού ΑΕ, δηλαδή αύξηση 1,6%. Και πάλι έχουμε ένα περιθώριο υγιές, δηλαδή 1,6 δισεκατομμύρια, που θα ενεργοποιηθεί αν χρειαστεί. Και έχουμε και το μηχανισμό ευελιξίας στις πληρωμές 45,7 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Και αυτή είναι η πίεση που προκύπτει κυρίως από το μεταναστευτικό. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού, ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες ε, που Στήριξτε και εσείς περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη, επενδύσεις, στήριξη της ανάκαμψης. Περίπου το, ο μισός προϋπολογισμός, ε, περίπου 66% πάνε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στον Ορίζοντα 2020, στο Συνδέοντο στην Ευρώπη, στην Ενεργειακή Ένωση, στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά και στην Πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση των νέων. Θέλουμε ο νέος προϋπολογισμός να διευρύνει και να εμβαθύνει την εσωτερική αγορά, γιατί γνωρίζουμε ότι η εσωτερική αγορά είναι η βασική πηγή της ανταγωνιστικότητάς μας. Δεύτερος, δεύτερη προτεραιότητα, να ανταποκριθούμε στις νέες εξελίξεις και να ενισχύσουμε γενικώ την Ευρώπη, να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές πιέσεις και το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει αύξηση, να ενισχύσουμε γενικώ στο, στο παγκόσμιο προσκήνιο την Ευρώπη και φυσικά χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, υγιή οικονομικά. Αυτό περιμένουν οι πολίτες, μη υπεύθυνη και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Και για τέταρτη συνεχή χρονιά συνεχίζουμε τη μείωση κατά 1% του προσωπικού. Και όπως γνωρίζετε και από προηγούμενες συνομιλίες που είχαμε, θα έχουμε και μια αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε με λιγότερους πόρους ε, να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Θέλουμε επίσης βιώσιμο προϋπολογισμό. Δαπανίσαμε άπειρες ώρες, εργόδεις προσπάθειες ε, ε, για τις πληρωμές, προκειμένου να προσαρμόσουμε τις νέες ε, αυτές αλλαγές στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και καταφέρνουμε επιτέλους ε, να έχουμε πιο βιώσιμο προϋπολογισμό. Τώρα, πού θα πάνε τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Γνωρίζω ότι είναι επώδυνοι αυτοί οι πίνακες. Σας έχουμε στείλει όμως το έγγραφο και βλέπετε την κατανομή και μάλιστα και τη σύγκριση με τον περσινό προϋπολογισμό. Αυτό που σας προτείνουμε είναι ε, η πληρώσεις, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ανακεφάλαιο και τη σύγκριση με το 2015. Και δεν είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια προσαρμογή γιατί το 2015 είχαμε τον διορθωτικό προϋπολογισμό 4. Οπότε εκεί η ανάληψη από τις, ε, στις αναλήψεις υποχρεώσεων είχαμε το 21,9 δις από το 2014. Είχαμε ένα επιπλέον πόσο. Πάντως σχεδόν, όλες τις, ε, σχεδόν όλα τα κεφάλαια έχουμε αύξηση και στις αναλήψεις υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών. Και αυτό με το ουδέτερο αναπρογραμματισμό. Στα θέματα της ε, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, για παράδειγμα, φαίνεται ότι στις αναλήψεις υποχρεώσεων ε, έχουμε μείωση 16%, αλλά στην ουσία έχουμε 3,5% αύξηση. Μετά τη διόρθωση που έγινε από την μεταφορά των 21 ε, δισεκατομμυρίων. Με παρακολουθείτε? Βλέπετε λοιπόν στο διορθωμένο πίνακα, στο κόκκινο, τι έγινε μετά από την ασυνήθιστη μεταφορά από το 2014 στο 2015 αναλήψεων υποχρεώσεων. Και μας μένει η πραγματική σύγκριση μεταξύ των προϋπολογισμών του 2015 και του 2016. Με απλά λόγια. έχουμε συνολικά αύξηση 2,4% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και 1,6% αύξηση της πιστώσεις πληρωμών. Βέβαια είναι αμελητές αυτές οι αυξήσεις, αλλά αν μη τι άλλο έχουμε πιο υγιή προϋπολογισμό. Νομίζω το πιο σημαντικό ακόμη είναι η επόμενη διαφάνεια. Α, συγγνώμη, ξέχασα τα περιθώρια. Εδώ βλέπετε τα περιθώρια που αφήσαμε και στις πληρωμές και στις αναλήψεις υποχρεώσεων. Θα θυμάστε ότι στις διαπραγματεύσεις για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς και του 2014 και του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την υποχρέωση να υποβάλει ένα συνετό προϋπολογισμό για το 2016 ώστε να μην εξαντλήσουμε από την αρχή τα περιθώρια και το καταφέραμε. Και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή σε όλες οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως αυτές που ασχολούνται με τα σημαντικότερα κεφάλαια και το πιο σοβαρό έργο. Και η επιμονή σας να βελτιώσουμε τις προβλέψεις μας, τις πληρωμές, αποδίδουν, γιατί τελικά καταλήξαμε σε πολύ πιο αξιόπιστες προοπτικές. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, πιστώσεις πληρωμών. Τι φαίνεται εδώ. Εδώ αποδεικνύουμε ότι βαίνουμε στο σωστό δρόμο με νέα προγράμματα που ξεκινούν και παλιά προγράμματα που σταδιακά κλείνουν. Είναι σημαντικό να γίνει αυτή η μετάβαση από τα παλιά στα νέα προγράμματα. Γιατί χωρίς αυτή τη μετάβαση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή γνωρίζουμε ότι θα καταλήξουμε και πάλι σε ένα σωρό ανεξόφλητων λογαριασμών που δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε. Έχουμε τώρα αύξηση 80% στις ε, πιστώσεις πληρωμών για τα νέα προγράμματα σε σχέση με το 2015. Οπότε το 2016 έχουμε 39% το μερίδιο των νέων προγραμμάτων, ενώ το 2015 ήταν 22 μόνο 100. Και συνεχίζουμε τις πιέσεις για συνετή και ορθολογική εκτέλεση των προγραμμάτων, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από τα παλιά στα νέα προγράμματα και να αποφύγουμε δυσάρεστο κλείσιμο της προηγούμενης περίοδου προγραμματισμού. Τώρα, διοικητικοί περιορισμοί και περικοπές στις διοικητικές δαπάνες. Βλέπετε τον πίνακα που αναφέρει τις διοικητικές δαπάνες ανά θεσμικό όργανο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αύξηση 1,5% Το Συμβούλιο έχει τη μικρότερη αύξηση και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σε μερικές περιπτώσεις είχαμε δικαιολογημένη αύξηση, όπως ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των δικαστών και στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είχαμε ε, πολλές κρίσεις ε, στις γειτονικές μας χώρες, γι' αυτό και δικαιολογημένα είχαμε αύξηση των δαπανών στην ΕΙΕΔ. Μάλιστα αποφασίσαμε να ανοίξουμε γραφεία και στο Ιράν, δεδομένης της κατάστασης ε, των διαπραγματεύσεων. Επίσης, ε, είπαμε ότι θα ανοίξουμε γραφεία και στο Μογκαντήσιο. το γραφείο είναι πολύ δαπανηρό εξαιτίας των επισφαλών συνθήκων ασφάλειας. Εξού και η μεγάλη αύξηση στην Ε.Ε. Πάντως ζητήσαμε από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να είναι πολύ προσεκτικό και να φροντίσει στο μέλλον να κάνει περικοπές και οικονομίες, ώστε αυτή η αύξηση να μην συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σε μερικούς οργανισμούς, το Frontex για παράδειγμα, ε, στον Οργανισμό για τη Μετανάστευση έχουμε εύλογες πιέσεις. Είναι πολιτική προτεραιότητα αυτό. Εξηγούνται έτσι μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτά και είναι αυτονόητο ότι θα είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν εγκρίνει αυτές τις διοικητικές περικοπές και τους περιορισμούς. Τώρα, Γνωρίζουμε ότι θα γίνουν οι αναγνώσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα γίνουν ενημερώσεις στη διάρκεια του έτους και μάλιστα έχουμε το παραδοσιακό, την παραδοσιακή διορθωτική επιστολή για τις γεωργικές δαπάνες. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τους τριμέρεις διαλόγους και τις ειδικέ διοργανικές συναντήσεις και θα τονίσω δύο τέτοιε συναντήσεις, μία για τους οργανισμούς, γιατί είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με τους οργανισμούς Είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να γίνουν ε, διεξοδικές αναλύσεις για τη διάρθρωση των, οργανισμών συγγνώμη, στις διάφορες κατηγορίες και στις ηθίκες. Για παράδειγμα, έχουμε οργανισμούς ε, που αυτοχρηματοδοτούνται, γιατί χρεώνουν τις υπηρεσίες τους. Οπότε τέτοιοι οργανισμοί θα έχουν μια φυσική ανάπτυξη που είναι διαφορετική ε, από αυτή των υπόλοιπων οργανισμών. Και παρόλα αυτά τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Αν θέλουμε κάποια μέτρα αποτελεσματικότητας για τους οργανισμούς αυτούς και μια αξιόπιστη διαδικασία για να διαχειριστούμε την ανάπτυξή τους, που είναι πιο φυσιολογική, και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία γι' αυτό. Επίσης έχουμε οργανισμούς που αναπτύσσονται λόγω εξωτερικών παραγόντων, οικονομικών όπως ο Οργανισμός για τη Μετανάστευση και Frontex. Εκεί θα πρέπει να υιοθετήσουμε διαφοροποιημένη προσέγγιση για τους διάφορους οργανισμούς. Πάντως, δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια λύση για όλους τους οργανισμούς, γιατί κάτι τέτοιο τεχνητά περιορίζει την ικανότητα των οργανισμών να μας εξυπηρετήσουν. Τώρα έκανα το λάθος να αναφερθώ σε κάτι που θα αποτελέσει το αντικείμενο των διοργανικών ε, συναντήσεων στο μέλλον. Και στα τέλη του φθινοπόρου θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις του προπολογισμού με την ε, περίοδο συνδιαλλαγής 29 Οκτωβρίου με 18 Νοεμβρίου. Εκεί θα βάλουμε τα δυνατά μας ώστε η περίοδος ε, συνδιαλλαγής να αξιοποιηθεί στο έπακρο, παραγωγικά, καθ' όλη τη διάρκειά της και όχι η τελευταία στιγμή, ώστε να ολοκληρώσουμε την απόφαση για τον προϋπολογισμό πριν χτυπήσει το ρολόι μεσάνυχτα στις 18 Νοεμβρίου. Αυτά και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να έρθω και να σας παρουσιάσω τον προϋπολογισμό. Και είναι εδώ και ο Σιλβάνο που θα απαντήσει σε πιο λεπτομεριακές ερωτήσεις αν διατυπωθούν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία μου, σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση την οποία αισθανθήκαμε ότι σε συγκινεί. Σας το ακούσαμε στη φωνή σας γιατί είναι ο πρώτος σας προπολογισμό. Αυτός είναι ο δικός σας προπολογισμό. Και είμαι βέβαιος ότι το φροντίσατε όσο του έπρεπε. Ε, σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για αυτή την παρουσίαση και κατανοώ ότι θα πρέπει να κάνετε διάφορες ανακοινώσεις αλλά θα μπορούσατε να μείνετε μέχρι τις 11. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε όλοι σύντομοι στις παρεμβάσεις μας. Άρα λοιπόν πρόκειται για έναν προπολογισμό ο οποίος στην ουσία αναλύει και το τον Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στατικικές Επενδύσεις κατ' ουσίαν και για τα υπόλοιπα ταμεία θα έχουμε άλλες ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάντες καταρχήν που είναι ο συντονιστής... Ε, ε σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Αντιπρόεδρο καταρχήν και θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο και όλους τους συναδέλφους καθώς και να συγχαρώ όλος ιδιαίτερο στον πρόεδρο της, Επιτροπή, της Επιτροπής είχαμε πολύ μακρόχρονες συνεδριάσεις ακριβώς λόγω του ΕΦΣΥ, του, στρατηγικού, του Ταμείου μάλλον Στρατηγικών Επενδύσεων και είμαστε έτοιμοι να προσπαθήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχόλια τα οποία κάνουμε κάθε χρόνο. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας περιορισμένος προπολογισμό ε, από τι ε, συνθήκες και από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ποτέ δεν θα είναι ένας τεράστιος προϋπολογισμός. Οι πληρωμές αντιστοιχούν μόλις το 1% του ΑΕΠ. 0,98 μάλιστα, ούτε καν 1% και επιπλέον και όσον αφορά τις υποχρεώσεις ανεβαίνει λίγο πάνω από το 1%, 1,0% σε σχέση με το ΑΕΠ. Αυτή η πρώτη φράση λοιπόν εξηγεί τον περιορισμό του προπολογισμού, αν θέλουμε να τον συγκρίνουμε με τον προπολογισμό των ΙΠΑ, που είναι 20% του εσωτερικού ακαθάριστου προϊόντο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικός προπολογισμό. Όχι, είναι σημαντικός και οι, πληρω... οι πληρωμές 143,5 δι ευρώ είναι κάτι το σημαντικό και γι' αυτό και είναι ε, ε, αυτό το σχέδιο τόσο σημαντικό. Εγώ λοιπόν εκφράζω την ικανοποίησή μου για αυτό το προπολογισμό που είναι ένας προπολογισμό επενδύσεων. Μόνο το 6% αφιερώνεται στις διοικητικές δαπάνες, το 24% είναι, ε, προορίζεται για επενδύσεις και για να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της, του Κοινοβουλίου. Έχουμε την απασχόληση της επιχειρήσης και κυρίως της μικρομεσαίες και έπειτα την ανάληψη ε, κινδύνου. Έχουμε λοιπόν αυτό που φαίνεται στην, στον τίτλο 1, όπου έχουμε τα διάφορα προγράμματα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και χαίρομαι για τις ε, τις υποχρεώσεις για αυτό το τίτλο, αλλά και για τις πληρωμές στον, στην κατηγορία 1α. Επίσης ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ε, εσωτερική αλληλεγγύη. Εσωτερική αλληλεγγύη ε, που είναι πολύ σημαντική. Η κατηγορία 1β που έχουμε πολύ σημαντική πολιτική που επίσης συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Χαίρομαι που εδώ έχουμε αύξηση όσον αφορά τις υποχρεώσεις. Και επίση ε, η πτυχή των ε, πληρωμών είναι αυξημένη σε σχέση με το 2005 και θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξαναδούμε αργότερα. Τώρα, οι άλλε προτεραιότητε και η εξωτερική αλληλεγγύη ε, ε, μας ικανοποιεί επίσης. Είμαστε στην τρίτη κατηγορία, ασφάλεια και ηθαγένεια. Έχουμε σημαντική αύξηση και εδώ. Και έχουμε επίσης αύξηση στην κατηγορία ε, Παγκόσμια Ευρώπη. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε την ανάγκη ε, που υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μην ξεχνά ποτέ την αλληλεγγύη. Στρεφόμενης και μετατρέποντας αυτή την αλληλεγγύη σε συγκεκριμένες δράσεις. Εδώ η συγκεκριμένη δράση που βλέπουμε είναι ο προϋπολογισμός στην τίτλο 3. Έχουμε 17,1% μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις και στην 3 και στην 4 έχουμε 28,5% και πράγμα που δείχνει ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει και αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη Μεσόγειο αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στη γειτονιά μας όπως αυτή, αυτό της Ουκρανίας. Για τα υπόλοιπα δεν έχουμε λεπτομέρειες και δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα αυτή τη στιγμή σε γραμμές και σε προγράμματα. Για να δούμε ακριβώ που υπάρχουν οι αυξήσει που γίνονται. Μάλλον οι αυξήσει δεν ξέρω τι γίνεται με το Frontex, με τα άλλα προγράμματα που σχετίζονται με όλους αυτούς τους τίτλους. Ε, θα χρειαστεί πιο εις βάθος και πιο λεπτομερής ανάλυση. Επίσης, ποιος είναι ο αντίκτυπος του πλάνου Juncker, του FSE, στον προϋπολογισμό, ε, θα το δούμε. Ελπίζω πως απόψε το βράδυ θα βρεθεί και μια συμφωνία για το FSC. Στην ε, στιγμή αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο που προέβησε λεπτομερή ανάλυση και γνωρίζοντα βέβαια πάντοτε πως οι περιορισμοί ε, για τον προπολογισμό είναι συγκεκριμένοι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ώστε οι υποχρεώσεις που αναλάβουμε στο πλαίσιο του PDP θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτούς και συγκεκριμένα για να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία ώστε αυτό ε, το, εδώ το κοινοβούλιο που δέχτηκε να εγκρίνει αυτό το πολιετές ε, ε, σχέδιο να μπορέσει να χρησιμοποιήσει στο έπακρο την ευελιξία και τα όργανα που του προσφέρονται, τα μέσα που του προσφέρονται και το Συμβούλιο να μπορέσει να ξαναθυμηθεί και διαρκώς εμείς θα πρέπει να θυμίζουμε στο Συμβούλιο τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει και που ανέλαβε σε αυτό το πλαίσιο και όλα όσα βρίσκονται στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο όσον αφορά τις υποχρεώσεις δηλαδή όλα όσα υπάρχουν εκεί δεν είναι τίποτα το νέο. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αναθεώρηση, πρόκειται για ε, ανηλυμένες υποχρεώσεις και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές. Πάκτα σουν σερβάντα. Δηλαδή οι ανηλυμένες υποχρεώσεις πρέπει να τηρούνται. Αυτό ξέρουν οι πολίτες και αυτή ακριβώς την πίστη έχει πάντοτε το Ευρωκοινοβούλιο και αυτό απαιτεί και από τους ε, εταίρους του. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεπρέ τώρα θα πάρει το λόγο, αν θέλει, ως εισηγητής των άλλων τμήματων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, περίμενα να είναι η σειρά της κυρίας Γκάρδια Ζαμπάλ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε την Πρόεδρε, επειδή αναφερθήκατε σε μένα. Εγώ δεν είμαι ε, ε απόλυτος στον προπολογισμό, αλλά ε, είμαι ε, πιστός στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ε, που θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σωστά, όπως πιστεύουν εξάλλου και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Τώρα, σε σχέση με το σχέδιο αυτό προπολογισμού, κυρία Αντιπρόεδρε, έγινε αναμφίβολα μεγάλη προσπάθεια και το λέω αυτό ότι ο πρώτος σας προϋπολογισμός είναι νέας ε, έκδοσης. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όμως. Καταρχήν για τα περιθώρια που, υπάρχουν, που παραμένουν διαθέσιμα, Ε, που αναφέρονται στις διαπραγματεύσεις που γίνονται σε σχέση με το Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων. Νομίζω πως υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμό πιο σημαντικό, το οποίο θα μπορούσαμε να δώσουμε για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, που ε, εξάλλου έχουν εκφραστεί εντόνως στις παράλληλες συζητήσεις που γίνονται για την ώρα. Να πω ότι για τις προτεραιότητες ε, του προπολογισμού για το 2016 ε, λέμε το ορίζοντας 2020 και το η διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Το παραθέτω με χιούμορ, όμως πιστεύω πως όταν είναι σκόπιμο να γίνει μια παραπάνω προσπάθεια, πως αυτά τα οποία γράφονται εδώ δηλαδή θα έπρεπε να συμφωνούν περισσότερο με το μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα για το προσωπικό ήδη εγώ Ήδη μάλλον το αναφέραμε και χθε, δηλαδή μείωση του 5%. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και ήδη έχουμε συζητήσει με κάποιους συνεργάτες σας. Μία μείωση που επηρεάζει το προσωπικό το οποίο είναι ε, τοποθετημένο στις αποστολές θα πρέπει να το κάνουν όλες, ε, όλα τα ιδρύματα, όλοι οι θεσμοί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κάνει επίσης. Αλλά αν έχετε νέες προτεραιότητες, ορισμένα θεσμικά όργανα έχουν περισσότερο περιθώριο αναδίπλωσης ε, δεδομένο του αριθμού των υπαλλήλων που έχουν, θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Να υπάρξει μια κάποια άλλη δηλαδή ευελιξία όσον αφορά τη μείωση του 5%. Μάλιστα ανοίξατε κάποια πόρτα που είναι χρήσιμη όσον αφορά τους διάφορους οργανισμούς. Θα είναι προς το συμφέρον μας όλα αυτά να τα δούμε πιο συγκεκριμένα στην επόμενή μας συζήτηση. Τίτλος 3. Ασφάλεια η κινητοποίηση των επιστώσεων είναι σημαντική σε σχέση με τους στόχους, γιατί αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 15 είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με τις πραγματικές περιστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέχρι το τέλος του έτους και κυρίως στις αρχές του επόμενου έτους. Το ίδιο και όσον αφορά το 4, τίτλο 4, ωστόσο θα ήθελα να πω κάποιες σκέψεις ε, σε σχέση με τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Είπατε ότι θα, αρχίσει, ότι θα ανοίξει μια αντιπροσωπεία σε Τεχεράνη. Δεδομένων των όσων μόλις έγιναν. Όμως θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή, αν είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Και πώς ε, θα μπορέσουμε να το στηρίξουμε. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αυτά που θέλω να πω και να επιφυλαχθώ για τα άλλα σχόλια και επικρίσεις μετά τη μελέτη εις βάθος του θέματος. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που δώσατε στήριξη στα όνειρα που, τρέφαμε μέχρι, που σήμερα το βράδυ, κύριε Φερνάνδης. ευχαριστώ σε εσάς, κύριε Αντιπρόεδρε. Εφόσον πρόκειται για τη σύσταση του Ταμείου Αγγίσεων για το ΕΦΣΥ. Κυρία Καρδία Ζαμπάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κρίμα που δεν μου δώσετε το λόγο πριν τον κύριο Ντεπρέ. Γιατί θα έπρεπε να... Δεν θα χρειαζόταν να μιλήσει καν, θα έλεγα και εγώ ακριβώς τα ίδια. Και εγώ σημείωσα τα περιθώρια, γιατί επειδή όλοι έχουμε στο μυαλό μας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, οπότε τα 2,2 δις σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να πάνε κάλλιστα και στο ταμείο αυτό το Εύση. Και δεν νομίζω ότι ιστορία το... στην ιστορία των, των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εξαντλήθηκε ουδέποτε ένα τέτοιο περιθώριο 2,2 δις. Οπότε θα μπορούσαμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το περιθώριο για να χρηματοδοτήσουμε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή άλλες πολιτικές μας προτεραιότητες. Γιατί εκεί που έχουμε τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις, συμπίπτουν απόλυτα οι προτεραιότητες αυτές με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ψηφίσαμε στους γενικούς μας προσανατολισμούς για τον προϋπολογισμό. Τώρα, πιο διεξοδικά, συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις ε, για το ΕΦΣΙ, για τον ορίζοντα 2020 και το συνδέοντα στην Ευρώπη. Το ορίζοντα 2020 και το συνδέοντα στην Ευρώπη είναι κατά κάποιο τρόπο τα θύματα του ΕΦΣΙ. Τώρα, για την πρωτοβουλία για τους νέους, για την απασχόληση των νέων, έχω κάποιες αμφιβολίες. Διάβασα το έγγραφο και δεν βλέπω τίποτα καινούριο στη δημοσιονομική γραμμή. Μηδέν ευρώ στις αναλήψεις υποχρεώσεων, αν δεν κάνω λάθος, για την πρωτοβουλία των νέων. Εκτός αν ε, εγώ παρέβλεψα κάτι. Και έχουμε και κάποιες πληρωμές που έχουν μεταφερθεί από πέρυσι και πρόπερσι. Δεν έχουμε τίποτα καινούριο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Οπότε να το αναφέρετε ως προτεραιότητα του 2016 μου φαίνεται υπερβολικό για να μην πω τίποτα πιο βαρύ. Φαντάζομαι ότι αυτό θα, θα είναι κάποιο λάθος που έγινε. Ελπίζω αυτά που αναφέρετε ως προτεραιότητες να έχουν και κάποιο δημοσιονομικό αντίκρισμα. Γιατί η μεταναστευτική πίεση, τα προγράμματα των κατηγοριών 3 και 4 ήταν ανέκαθεν προτεραιότητα και ήταν και τα πιο σημαντικά κεφάλαια που μάλιστα ιστορικά υποχρηματοδοτούνταν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Έχουμε τώρα κάποιες αυξήσεις, μάλιστα ακόμη και 12% σε μερικά κεφάλαια, πολύ σημαντικό πρόοδος, αλλά να δούμε και τις λεπτομέρειες, ώστε να εξακριβώσουμε αν όντως οι πολιτικές προτεραιότητες έχουν αντίκρισμα και στα, στους αριθμούς. Γιατί αν δεν υπάρχει τέτοιο αντίκρισμα και τέτοια ανταπόκριση, δεν κάνουμε προπολογισμό, αλλά marketing. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, να προσδιορίσουμε όλα τα ποσά και να δούμε πώς θα επηρεάσει το ΕΦΣΙ τον ορίζοντα 2020 και το συνδέοντα στην Ευρώπη, για να διορθώσουμε με την δημοσιονομική διαδικασία κάποιες περικοπές που έχουν προβλεφθεί. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κορδιά Σάμπαλ. Συνεχίζουμε με τους συντονιστές. Η κυρία Μυριάντα. Ε, ο κύριος Τόμ. Α, ο κύριος Άσχορθ που αντικαθιστά το συντονιστή. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας παρουσιάσατε τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να πω που, ότι με έχει ενθαρρύνει πάρα πολύ το γεγονός ότι κάνατε δύο σχόλια στο τέλος της παρουσίασής σας. Είπατε καλύτερη εστίαση και καλύτερη πειθαρχία. Αυτό πραγματικά με ευχαριστεί ιδιαίτερω και αυτό ακριβώς θα θέλαμε να δούμε. Αυτό περιμένουμε άλλωστε και από εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τα θέματα εστίασης. Έχετε φιλοδοξία να κάνουμε πιο πολλά με πιο λίγα χρήματα. Πολύ σωστά. Θαυμάζω το γεγονός ότι ανταποκριθήκατε στις ε, τρέχουσες προκλήσεις, απασχόληση, μετανάστευση. Ουκρανία, ήσασταν ρεαλιστικοί στην παρουσίασή σας. Θα πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες βέβαια, είναι φέτο χρόνο. Και προσβλέπω στη συζήτηση του πώς μπορούμε να κοιτάξουμε τα πιο ασθενή σημεία, όπως για παράδειγμα τις υπηρεσίες, όπως αναφέρατε και εσείς ίδια. Σε θέματα πειταρχίας τώρα. Καλωσορίζω επίσης τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας για τις απλήρωτους λογαριασμούς. Ο στόχος των 2 εκατομμυρίων μέχρι τα τέλη του 2016 είναι αισιόδοξη πρόκληση. Καλή τύχη σας εύχομαι. Η ζωή δυστυχώς δεν είναι πάντα τόσο εύκολη και πολύ φαντάζομαι, πολύ ε, υποπτεύομαι μάλλον ότι θα είναι δύσκολο να το πετύχετε. Αλλά θαυμάζω την φιλοδοξία σας. Χρειαζόμαστε φιλοδοξία. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να θέσω εξακολουθούμε να έχουμε το πρόβλημα των ράλς βέβαια. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Τα μέλη της Επιτροπής θα ήθελα να ακούσουν ποιο είναι το βιώσιμο επίπεδο ράλ. Και αν θα θέλατε να μας πείτε πώς προβλέπετε ότι θα διακυμανθεί το επίπεδο αυτό στο μέλλον. Να τονίζω την ανάγκη να εμπλακούν πιο πολύ τα κρατημέλη. Γιατί για να δεχτούν την πειθαρχία και τη συνεργασία τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια μεγάλη προτεραιότητα για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Καλώς ορίζω το σχόλιο για τα περιθώρια. Είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι για το ΕΦΣΥ, για το Ταμείο Επενδύσεων, αλλά ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και τέλος, με πολύ ευγενικό τρόπο μας είπατε το εξής ο έλεγχο των διοικητικών εξόδων των θεσμικών οργάνων. Θεωρώ ότι αυτό με πολύ τακτικό τρόπο λέει στο Κοινοβούλιο αν τα πετυχαίνουν αυτές τις μειώσεις τα άλλα θεσμικά όργανα γιατί έχει το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Επίτροπε, θέλουμε όντως καλύτερη εστίαση και καλύτερη. Σας ευχαριστώ, κυρία Ευχαριστώ. Νομίζω πως όλοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές ε, αλλά θα πρέπει να το μελετήσουμε εις βάθος για τα ειδικά μέσα όταν ε, μιλάτε τι, ποια είναι αυτά και έπειτα βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην αλληλεία και γεωργία και στην φυσική ζωή. Αυτές τις λεπτομέρειες ε, νομίζω θα πρέπει να βάλουμε να λείπουν και συμμερίζομαι ε, σε σχέση με ε, τις ανησυχίες για το σχέδιο Juncker. Θα καλύψει το κενό που έχει αφήσει το Connecting Europe και, το, και, και η έρευνα και η ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Όπως ακούσατε ήδη, όλοι οι συνάδελφοι προτίθεται να σας συγχαρούν για τις εξαιρετικές προτάσεις σας για τον ε, προπολογισμό του επόμενου έτους. Τι να κάνω κι εγώ, θα συμφωνήσω μαζί τους. Τρεις μικρές παρατηρήσεις ωστόσο. Ερωτηματικά, σχόλια, παρατηρήσεις, όπως θέλετε πείτε το. Δεν άκουσα, δεν ξέρω αν φταίω εγώ. Είπατε ότι πρέπει να πρασινίσει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το κάνουμε αυτό. Τι σημαίνει αυτό κατελάχιστον. Κοιτώντας τα αριθμητικά στοιχεία για, την, ε, το ίτερ, για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στην Γαλλία. η μείωση αυτού θα με ικανοποιούσε. Ένα άλλο θέμα που θα Έλπιζα να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε γιατί δεν το καταλαβαίνω εις βάθος. Είναι αυτό το στρατηγικό ταμείο επενδύσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016. Πώς ε, συνδυάζονται ακριβώς, όπως είπε και ο κ. Σάσουαρτ. Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε πιο πολλά με πιο λίγα χρήματα. Και τρίτον, αν κατάλαβα και πάλι καλά, Σε ό,τι αφορά την ε, αντίδραση στις πιέσεις τις μεταναστευτικές, σκοπεύουμε να δαπανίσουμε χρήματα με έναν ανισόρροπο λίγο τρόπο. Η υπεύθυνη ασφάλεια θα είναι αρκετά ικανοποιημένη από αυτά που τους προτείνουμε. Αλλά τα ποσά για την νόμιμη μετανάστευση φαίνεται ότι μειώνονται. Ε, ε, έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. γιατί οι σύμβουλοι μου καταρτίζουν σχετικού πίνακε, καταλαβαίνετε. Αν αυτό δεν αληθεύει, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτή είναι η εντύπωση που έχω σχηματίσει έω τώρα. Γιατί αν όντω ισχύει αυτή η προσέγγιση, θα ήταν πραγματικά άσχημη η κατάσταση, σχολιάζει η κυρία Χολμαέρα, αλλά εκτό μικροφώνου. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαι κάπω. Ε, έκπληκτος, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το τι σημαίνουν τα αριθμητικά στοιχεία αυτά, αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι πρόκειται να τα ε, εξηγήσουμε. Ο κύριος Γκάιερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Γεωργιεβά που μας παρουσιάσατε τα πιο σημαντικά στοιχεία του προπολογισμού του επόμενου έτος. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω για τα αριθμητικά στοιχεία αυτά και κάποια σχόλια από δικής πλευράς επίσης στη σελίδα 6 και 7. Εξ όσων το κείμενο και από ότι τονίσατε το κόκκινο τμήμα στη σελίδα 7 τα καθοριστικά αριθμητικά στοιχεία είναι αυτά που συνεπάγονται από τον προπολογισμό του 2015, του τρέχοντος έτους. Οι υποχρεώσεις ε, από το 2014 μια περίπτωση που εμφανίστηκε μία φορά και αν το υπολογίσουμε έχουμε 2,4% αύξηση στις υποχρεώσεις, 2,6% αύξηση στις ε, πληρωμές. Αλλά μιλάμε για 10 εκατομμύρια. Και είναι σημαντικό να σχολιάσετε Πώς ε, σχετίζεται αυτό στο γενικότερο πρόβλημα των ποσών υπόλοιπου προς ακαθάριση. Κοιτώντας λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία αυτά, έχουμε λοιπόν ε, δέκα δις διαφορά μεταξύ των πληρωμών και των δεσμεύσεων. Μήπως μειώνεται αυτό το κενό πολύ λιγότερο από ό,τι θα μπορούσε να μειωθεί. Θέλουμε μια πολιτική βάση αριθμητικών στοιχείων. Και αν πάρουμε αυτή τη βάση, η αύξηση του προπολογισμού στο τομείς 3 και 4 στην ασφάλεια και σε τομείς όπως ε, το Global Europe είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο, είναι σωστή. Το επόμενο βήμα είναι να συμφωνήσει και το Συμβούλιο για τα αριθμητικά στοιχεία αυτά. Και εμένα με απασχολούν δύο πράγματα. Κατά πόσον θα θυμηθεί τη δέσμευση του το Συμβούλιο για την επίλυση της ε, κρίσης των πληρωμών. Γιατί τα έχουμε συνηθίσει αυτά από το Συμβούλιο. Δεσμεύσεις οι οποίες ε, μετά από 24 ώρες ε, με διαφορετικό μορφότυπο εγκαταλείπονται. Θα ήθελα να προειδοποιήσω το Συμβούλιο γιατί αν ισχύουν όλα όσα συζητήσαμε για την κρίση των πληρωμών και σε ό,τι αφορά τις ιδιαίτερες προκλήσεις, ε, τις πολιτικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα έτη, το Συμβούλιο δεν μπορεί να αρχίσει να διαγράφει και να μειώνει ποσά σε όλες τις κατηγορίες, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Άρα, μετά τις χθεσινές διαπραγματεύσεις, ε, Αναρωτιέμαι, όταν θα εξετάσει το, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά πόσο το Συμβούλιο θα θυμηθεί όλα όσα συμφωνήσαμε και συζητήσαμε για την κρίση πληρωμών. Κατά πόσο θα ακολουθήσει την παράδοση των τελευταίων ετών ή κατά πόσο θα λάβει υπόψη την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμεί από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προσέξουμε ιδιαίτερα το τι θα συμβεί. Χαίρομαι επίση, ε, ιδιαίτερω κυρία Γεωργεβά, για όσα είπατε για τι υπηρεσίε. Θα υποστηρίξω την, την προσέγγιση ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως το παρελθόν. Να διευκρινίσω και στους συναδέλφους ότι υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από τους οικονομικούς και βιομηχανικούς κλάδους. Έχουν έσοδα λοιπόν και παρέχουν μια υπηρεσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών που χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό κλάδο δεν μπορεί να έχει συμμεταχείριση με το προσωπικό άλλων τέτοιων υπηρεσιών. Θα λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτή την ε, διευκρίνηση για τις ε, υπηρεσίες. Ο κύριος Άσχορτ μίλησε για τα δύναμα σημεία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Ελπίζω ότι το ίδιο να εννοείτε και εσείς σας υποστορίζω σε ό,τι αφορά τα θέματα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προϋπολογισμού. Αν κοιτάξετε τον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, θα δείτε που είναι τα προβλήματα αυτά. Τα πιο πολλά προβλήματα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα μέτρα δεν ε, λειτουργούν επαρκώς σύμφωνα με την ανάλυση του, της Επιτροπής. Και θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση πραγματικά να διαμορφώσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τον προπολογισμό του και θα θέλαμε να ακούσουμε σχόλια και από τον Εμένα Βασίλειο. Η κυρία Γεωργίευα πρέπει στις 11 και 10, 11 και 4 το αργότερο να αποχωρήσει. Και έχουμε και τέσσερις ακόμη ομιλητές αν ε, θέλουν να προλάβουν να υποβάλουν τις ερωτήσεις και να ακούσουν και απαντήσεις, θα πρέπει να είναι πολύ λακωνικοί. Ο κύριος Μάνικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου αρκεί και ένα λεπτό. Το προπολογισμό ε, πιστεύω ότι ακολουθεί τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις ε, τρέχουσες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κυρία Αντιπρόεδρε, που ε, κάνετε προσπάθειες για τη μείωση των δεσμεύσεων το 2016. Πιστεύω ότι πραγματικά θα είναι καθοριστικό το έτος αυτό. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει στρατηγική που θα αποτρέψει την επανάληψη της ίδιας κατάστασης σε πέντε χρόνια. Στην παρούσα φάση είναι δυνατόν να μειωθούν οι δεσμεύσεις, αλλά σε πέντε έτη θα βρεθούμε σε μια παρόμοια κατάσταση ενδεχομένως. Υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική η οποία θα απέτρεπε την επανάληψη της κατάστασης σε ό,τι αφορά τις απειλωτές δεσμεύσεις, η κυρία uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα συμφωνήσω όσα υπόθηκαν για το ότι καλωσορίζουμε τη γενικότερη κατεύθυνση του προϋπολογισμού όπως παρουσιάζεται και σε ό,τι αφορά την πλευρά των πληρωμών στο 1α. Πολύ υποπτεύομαι ότι ο διάολος θα είναι στις λεπτομέρειες πέρα από την όλη συζήτηση που γίνεται για το ΕΦΣΥ Ελπίζω να υπάρξει έμφαση και στην επένδυση στην έρευνα. Πέρα από τους τομείς που θα προκαλέσουν μόχλευση. Μια απλή ερώτηση τώρα. Στο κεφάλαιο 3, σας διαφορά το περιθώριο. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό και θα συμφωνήσω με τα όσα υπόθηκαν επίσης και για τις υπηρεσίες. Θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω την διαφοροποιημένη μεταχείρισή τους. Ευχαριστώ κύριε Νόβακοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Να σας συγχαρώ, όχι όμως μόνο για τις προσπάθειες για το 2016, αλλά και για κάτι ακόμα γιατί κρίνοντας από την παρουσίαση ο προϋπολογισμός του 2016 στρίζεται πιο πολύ στα αποτελέσματα και όχι στα ποσοστά και στα αριθμητικά στοιχεία. Σας συγχαίρω. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, ε, εκατομμύρια ε, ευρωπαϊκές οικογένειες και όχι για αριθμούς. Να σας συγχαρώ για τις εγγύησεις, για τη νεολαία. Ε, γιατί είναι 7 εκατομμύρια και παραπάνω οι νέοι που ψάχνουν μια δουλειά. Και να σας δείσω μια χάρη στο κεφάλαιο αυτό. Συντονιστείτε καλά με την Επίτροπο Ταΐσεν, που είναι η συναρμόδια συνάδελφός σας. Προκειμένου να υπάρχουν τα χρήματα αυτά όταν θα χρειαστούν για τους νέους. Τέλος ο προϋπολογισμός διαβάζοντας ε, τις ε, λεπτομέρειες βλέπω ότι να είμαστε μικροί για τα μικρά προβλήματα και μεγάλοι στην αντιμετωπισή μας για τα μεγάλα προβλήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Merci. Σας ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Χολμάιρ είναι η τελευταία μιλήτρια. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι ειλικρινής και θα πρέπει να είμαι και σύντομη και αυτό θα με ξεκάθαρη. Έχω την αίσθηση ε, ότι το έγγραφο μας κρύβει κάποια πράγματα. Πιο πολλά μάλλον κρύβει παρά αυτά που λέει. Είχαμε στο παρελθόν παρουσιάσεις με τις στήλε, τι είναι αρνητικό, τι είναι θετικό. Στην περίπτωση όμως αυτή βλέπουμε μία παρουσίαση η οποία πιο πολλά ερωτηματικά δημιουργεί παρά απαντάει. Όπως ο συνάδελφο Γκάιερ για το θέμα των υπηρεσιών. Έχουμε υπηρεσίες όπου υπάρχουν ε, ανάγκη μεγάλε αλλαγέ Θα έχει την τόλμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τι μεγάλε αλλαγέ προσωπικού και σε ό,τι αφορά τις μεγάλες αλλαγέ στη χρηματοδότηση σε υπηρεσίε. Γιατί αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν ε, δίνει, δείχνει ότι ε, πολλά είναι τα μεγάλα και ωραία λόγια, αλλά δεν υπάρχει συνεπής ε, δράση και ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την έναρξη των προγραμμάτων, δεύτερο στοιχείο. Αυτό το διτυπώσαμε ξεκάθαρα στην προηγούμενη διαπραγμάτευση ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει καθυστέρηση της εκκίνησης των έργων. Τώρα βλέπουμε δύο χρόνια καθυστέρηση. Δεν θα έχουμε πιο λίγα κενά μεταξύ δεσμεύσεων και πληρωμών. Γιατί αν περνάνε δύο χρόνια μέχρι να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα χρειάζεται χρηματοδότηση δηλαδή τα δύο χρόνια. Και το πρόβλημα θα εμφανιστεί σε κάποια χρόνια. Είμαι δύσπιστη. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που μας προτείνεται αυτή τη στιγμή. Ή θα μειώσουμε τις αναλήψεις υποχρεώσεων ή πρέπει να βρούμε φρέσκο χρήμα. Νομίζω ότι συνεχίζεται λίγο το παιχνίδι, αλλά με πιο κομψή παρουσίαση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το δούμε αυτό στο τελική ανάλυση. Τι κρύβεται πίσω από τα αριθμητικά στοιχεία. Γιατί τα αριθμητικά στοιχεία και η παρουσίαση αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής, μου προκαλεί πιο πολλά ερωτηματικά παρά μου απαντάει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κανένα θαύμα για τις πληρωμές όταν ψηφίζουμε με τα δύο δισεκατομμύρια διαφορά στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, ουσιαστικά ε, αυξάνουμε τα ραλ, τα υπόλοιπα προς εκαθάριση και σκάβουμε το λάκκο μας όλο και πιο βαθύ. Κύριε Επίτροπε, οι εκτιμήσεις ήταν ε, εν γέννη πολύ θετικές και επικοδομητικές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και θα έχουμε πολλές ευκαιρίες ε, να συνεχίσουμε να βαθύνουμε στην ε, ανάλυση των ε, αριθμών. Σίγουρα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το θέμα των λεπτομεριών. Για ειδικέ ερωτήσεις που υποβάλλετε θα σας στείλω γραπτό στις απαντήσεις για να υπάρξει σαφήνεια. Τώρα, για κάποια γενικά μηνύματα να κάνω κάποια σχόλια. Ποια ήταν τα γενικά μηνύματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε μεγάλοι στα μεγάλα και πιο διακριτικοί στα θέματα ίσονος σημασίας. Και αυτό είναι δύσκολο, δύσκολο έργο να εντοπίσουμε κάποιες αρνητικές προτεραιότητες μετά από πολλές δεκαετίες που δεν ήταν απαραίτητο, δεν είναι και εύκολο. Πάντως προσπαθούμε να είμαστε σαφείς και να ε, καθοδηγούμαστε κυρίως από την ανάγκη να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας και κυρίως αυτούς που εξαρτώνται από εμά για να κάνουν σωστές επιλογές, είτε γιατί είναι άνεργοι, είτε γιατί έχουν τεράστια προβλήματα, είτε γιατί οι ερευνητές με φαϊνές ιδέες αντί να τις εφαρμόζουν και να τις διαθέτουν στην ευρωπαϊκή οικονομία φεύγουν, ξενιτεύονται και τις αξιοποιούν αλλού. Γι' αυτό και λέμε προτεραιότητα μας είναι να χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό το στόχο της εξυπηρέτησης του πολίτη τον προϋπολογισμό. Γιατί είναι μικρός αλλά θαυματουργός αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Ε, φυσικά δεν είναι κάτι που θα γίνει εν μία νυχτή ούτε ένα έργο που θα ολοκληρώσουμε με ένα προπολογισμό, αλλά σίγουρα αυτό είναι ο σκοπός και θα δουλεύουμε προς την υλοποίησή του. Κάποια επιμέρους σχόλια τώρα. Για τα περιθώρια. Τα περιθώρια έχουν λόγο ύπαρξης. Ε, μας επιτρέπουν να προσαρμοστούμε. Και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είπαμε ότι από τη στιγμή που θα αποσαφινιστούν τα περιθώρια του 2016 θα προσφέρουμε τη σαφήνεια αυτή για τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να μειώσουμε τις μεταφορές από τα δύο προγράμματα που θα χρηματοδοτήσουν μέρη το ΕΦΣΥ. Και αυτό κάναμε και πέρυσι. Ε, παροτρύνουμε το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται τέτοια παρότριση, να εξετάσει το κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και περισσότερο τα περιθώρια, αν το κρίνουμε απαραίτητο. Και μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για τα περιθώρια, χωρίς να διαταράξουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πώς θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να συνεχιστεί το επικοδομητικό πνεύμα και κλίμα μεταξύ των θεσμικών οργάνων και να καταλήξουμε σε καλή συμφωνία. Βέβαια, το σχέδιο του Juncker δεν είναι να το αντιμετωπίζουμε σε αντιπαράθεση με την καινοτομία ή το συνδέοντα στην Ευρώπη. Ίσα ίσα το σχέδιο Juncker θα στηρίξει και την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη και την έρευνα και την διασύνδεση των υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ψηφιακή οικονομία και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Τώρα, λέτε, μπορούμε όντως να θεωρούμε προτεραιότητα την πρωτοβουλία για τους νέους αν έχουμε μόνο πληρωμές και καμία ανάλυση υποχρεώσεων. Η απάντηση είναι καταφατική και ήταν συνειδητή η επιλογή μας να επιταχύνουμε τις αναλήψεις υποχρεώσεων ώστε να δημιουργήσουμε μία όθηση. Και το 2016 επικεντρωνόμαστε στις πληρωμές. Και έβαλα και την υπογραφή μου εδώ και συμφωνήσαμε για σημαντική προχρηματοδότηση της ε, πρωτοβουλίας για την ε, καταπολέμηση ενεργείας των νέων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πατήσουμε γκάζι και να επιταχύνουμε το ρυθμό μας. Έχουμε και την ενδιάμεση αναθεώρηση. Και στην ενδιάμεση αναθεώρηση θα εξετάσουμε τα περιθώρια και πού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αν στην ενδιάμεση αναθεώρηση Έχουμε την αίσθηση ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση η πρωτοβουλία για τους νέους. Ελπίζω να έχω, δείξουμε την πολιτική βούληση και να δημιουργήσουμε συνένεση, να συγκεντρώσουμε συνένεση για να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Πάντως έχω την αίσθηση ότι η πρωτοβουλία για τους νέους είναι προτεραιότητα και του προϋπολογισμού του 2016. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το πρασίνισμα του προϋπολογισμού. Συγγνώμη που το παρέλεψα, πώς συνέβη κάτι τέτοιο. Όντω είναι στόχο μα το πρασίνισμα, 20% του προπολογισμού να πάει στο πρασίνισμα, ε, η ειδική μνήμα στι κλιματικέ αλλαγέ. Εγώ θα προτιμούσα να είμαστε πάνω από 20%. Θα πρέπει να ε, μην φυστούμε προσπαθειών ώστε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο, το πρασίνισμα, που είναι σημαντικό για την οικονομία και το μέλλον μα. Για τα ράλς, τα υπόλοιπα προ εκαθάριση. Φυσικά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα της καλύτερης αντίληψης, καλύτερης διαχείρισης ε, των ΡΑΛ. Έχουμε διαφορά δεκαδείς αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό, ότι με καλή διαχείριση των νέων προγραμμάτων που ξεκινούν, που δρομολογούνται και είπατε γιατί καθυστερήσαμε τόσο γνωρίζουμε ότι 80% των ε, κονδυλίων είναι συνυπευθυνότητα κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το, κανδό, για το ταγκό χρειάζονται δύο παρτενέρ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και για τις προβλέψεις ε, των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών, ώστε όταν αυξάνουμε τις αναλήψεις υποχρεώσεων να ξέρουμε πώς θα τις χρηματοδοτήσουμε με τις πληρωμές που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Επίσης, να δούμε την πρόοδο κάποια στιγμή και σίγουρα θα πρέπει να κρίνουμε. Μπορούμε να κρατήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς με βιώσιμο τρόπο. Θα έχουμε καταρχήν την ενδιάμεση αναθεώρηση, το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί, με βάση τεκμήρια και αυτές αποδείξεις και αποδεδειγμένη χρηστή διαχείριση θα έχουμε περισσότερα εργαλεία για να δούμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε το έργο με τα κράτη-μέλη, όπως είπατε πολύ, ώστε και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν το δικό τους μέρος ευθύνης και να μην στέλνουν απλώς πληροφορίες, αλλά να διαχειρίζονται τα σχέδια, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες τους με συνετό τρόπο για να χειριστούμε καλύτερα τα ραλ και να μην ξεφύγουν από τον έλεγχό μας με αρνητικέ συνέπειες. Για τους οργανισμούς. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά και να λάβουμε απόφαση. Και αυτό θα γίνει στην διοργανική ομάδα για τους οργανισμούς. Αλλά επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Τι γίνεται ε, όταν έχουμε ε, ρήτρε ε, σταδιακής διακοπής sunset closes για τους οργανισμούς. Πού πηγαίνουμε με τέτοιες ρήτρε, πουθενά. Έτσι μόνο θα συνεχίσουμε. Μόνο σε μία περίπτωση είχαμε μία, ένα οργανισμό που διεκπαιρέωσε το έργο του. Οπότε το θέμα είναι, συνεχίζει να λειτουργεί, παρόλο που έχει ολοκληρώσει το σκοπό του. Ναι, η απάντηση είναι ότι ακόμη λειτουργεί, είναι ανοιχτή, ανοιχτός οργανισμός και λειτουργεί. Θα πρέπει να κρίνουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των οργανισμών με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Πρέπει να έχουμε τα κότσια, όχι απλώς την ικανότητα, τα κότσια, να κάνουμε την αξιολόγηση και να την συνοδεύσουμε με δράσεις. Γιατί ακόμη και όταν κρίνουμε ότι ένας οργανισμός δεν χρειάζεται πια, εξακολουθεί να είναι εν ενεργεία. Θα πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί με αυτά που δημιουργούμε, γιατί από τη στιγμή που τα ιδρύουμε, τα δημιουργούμε, θα παραμείνουν ε, ατέρμονα, ακόμη και αν ο σκοπός τους έχει εκλείψει. Ε, αν έχουμε σωστούς δείκτες αποδοτικότητας και τους εφαρμόζουμε αυστηρά με πυγμή και συνετά, με συνέπεια, μπορούμε να κρίνουμε τι θα πρέπει να συνεχιστεί και τι θα πρέπει να κλείσει. Μέχρι στιγμής δεν, ήμασταν, δεν είχαμε τα κόσια να, από πολιτική άποψη να προβούμε σε αυτή την κρίση. Ορίστε. Καλό θέμα αυτό για τη διοργανική ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Πάλι παρασύρθηκα. Βλέπετε ότι ασχολήθηκα πολύ με το θέμα αυτό τον τελευταίο καιρό. Και αυτό το λάθος έκανα και πριν, να συνδέω το θέμα των οργανισμών με την υπόλοιπη συζήτηση, ενώ είναι θέμα της διοργανικής ομάδας. Και μία ερώτηση για το μηχανισμό ευελιξίας, τους μηχανισμούς ευελιξίας. Είναι το αποθεματικό της κρίσης, το, το Ταμείο Αλληλεγγύης, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θεωρούμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί ευελιξίας βρίσκονται υπεράνω των ανώτατων ορίων. Έτσι τους αντιμετωπίζουμε. Βέβαια εδώ υπάρχει διάσταση απόψε με το Συμβούλιο παλιά και έχουμε και τρεις νέους μηχανισμούς. Το μηχανισμό ευελιξίας, το γενικό ε, περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και το αποθεματικό εκτάκτο ανάγκης. Και για τους σπόρους ε, θα σας στείλουμε τις λεπτομέρειες γιατί πρέπει να εξετάσουμε μεμονωμένα και διεξοδικά τα κεφάλαια. Θέλουμε πάντως ένα χρηστό υγιή προϋπολογισμό και να τον εφαρμόσουμε με συνετό τρόπο. Ελπίζω να μην παρέλειψα κάτι σημαντικό. Είπατε ότι ποτέ δεν είχαμε περιθώριο πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια. Το 2008 το περιθώριο ήταν 3 δισεκατομμύρια, σας πληροφορώ. Οπότε είχαμε μια περίπτωση στο παρελθόν με υψηλότερο περιθώριο. Πάντως εγώ για τα περιθώρια δεν είμαι υπέρ των μεγάλων περιθωρίων, μόνο και μόνο ως αυτό σκοπό. Θέλω υγιή περιθώρια, ώστε να μπορέσουμε όταν χρειαστούμε να κάνουμε τις προσαρμογές έχουμε το γενικό περιθώριο για πληρωμές και αναλήψη υποχρεώσεων και θα το συζητήσουμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Ό,τι δεν χρησιμοποιήσουμε θα το χάσουμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Αυτά και σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Και τώρα πραγματικά πρέπει να φύγω, να σταματήσω. Σας ευχαριστούμε κυρία Γεωργίευα. Θα δούμε τι υποδοχή θα επιφυλάξει το σχέδιο προϋπολογισμού σας στο Συμβούλιο. Και θα σας ενημερώσουμε τις επόμενες εβδομάδες για τις προτεραιότητες μας. Επιμείνατε στο θέμα της απασχόλησης των νέων. Είναι ένα θέμα που μιλά στους Ευρωπαίους. Αν όμως ε, θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις ε, για να δώσουμε ξανά την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στους νέους Ευρωπαίους που σήμερα είναι δίχως δουλειά, θα πρέπει να χρειαστεί μια δράση, πιστεύω, για την κινητικότητα. Και θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για το έρασμος και το έρασμος συν. Σας ευχαριστώ ε, είναι μικρός προϋπολογισμός, είναι επειδή είναι μόνο το 1% του ΑΕΠ και γι' αυτό και πρέπει να το προσέξουμε όλος ιδιαίτερος για να μπούμε στην ουσία και έπειτα θα μπορέσουμε με το δικό μας τρόπο να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Ευχαριστώ πολύ για την πολλά υποσχόμενη παρουσίασή σας. Merci, beaucoup. ce soir. Θα τα πούμε το βράδυ στον τριμερή για το FC που ελπίζω ότι θα είναι και ο τελευταίος. Ε, στα διάφορα έχει κανείς να μας πει κάτι. Όχι. Επόμενη συνεδρίαση 8 Ιουνίου στις 7. 7 με 9 το βράδυ στο Στρασβούργο. Χαίρετε. Πέρα συνεδρίαση.